Έχω λάβει ένα αίτημα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την ε, πρόταση διορισμών σε μια αντιπροσωπεία. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση μέχρι το τέλος συνεδρίασης,